Pan przewodniczący! Good afternoon. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε και πάλι την συνεδρίαση Έχετε λάβει τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Ως εκ τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια μας διάταξη των είναι δήλωση επιτροπής ως προς την έγκριση των τροποποίησεων της συνθήκης και θα ήθελα να επισημάνω στους κυρίες και κύριους βουλευτές ότι κατά την ε, συνεδρίαση αυτή δεν προβλέπεται, το τμήμα αυτό της συνεδριάσεως δεν προβλέπεται διαδικασία catch the eye, ούτε ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Ε, αναγνωρίζουμε όμως τη σημασία του θέματος και γι' αυτό το ε, χειριζόμαστε ως ζήτημα προτεραιότητας. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόν. Κύριε Πρόεδρε, Ζωσέ Μανουέλ Βαρόσο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα ε, θετική γνώμη ως προς την απόφαση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον προηγούμενο Δεκέμβριο για μια περιορισμένη τροποποίηση ε, του άρθρου 136 συνθήκης προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, στόχος είναι να επιτραπεί στα κράτη-μέλη με ε, νόμισμα το ευρώ, η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού που θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα, τη δημοσιονομική σταθερότητα του ευρώ στη ζώνη του ευρώ ολόκληρη. Και έτσι το 2013 θα αντικατασταθούν τα τωρινά προσωπικά μέσα, δηλαδή το ταμείο και ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα μέσα. Πρόκειται για μια απόφαση απαραίτητη για να επιβεβαιωθεί και η βούλησή μας να προσπιστούμε το κοινό μα νόμισμα και να εγγυηθούμε επί τη ουσία τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ε, εναντί των ανισορροπιών ορισμένων κρατών μελών στα δημοσιονομικά τους που πρέπει να αντισταθμιστούν και έτσι πρέπει να συμπληρωθεί σχετικά το πλαίσιο το ρυθμιστικό της συνθήκης. Πλην όμω, και όπω υπογράψα και εγώ στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάθε πρωτοβουλία μέσα στην, ε, στο πνεύμα τη ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση των ευρωπαϊκών ε, οικονομιών και υπογραμμίζω ανταγωνιστικότητα και σύγκληση των οικονομιών μας. Κάθε λοιπόν τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πνεύμα του σεβασμού τη συνθήκη και των αρχών και ρυθμίσεων, κανόνων που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία αυτή και των θεσμικών τη οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω εκ τούτου θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία νομοθετική ή άλλη έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εγγύηση τη συνοχή αυτού του μηχανισμού χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται σεβαστή η συνθήκη. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2011 με δήλωση αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού για τη σύγκληση στην ζώνη ευρώ για 17 κράτη-μέλη ε, και φυσικά για τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να ισχύσουν όλες οι διατάξεις της συνθήκης περί αρμοδιότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της και συγκεκριμένα περί των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αναφέρει ρητά με στη δήλωσή της 4ης ε, Φεβρουαρίου. Σήμερα με συζητούμε ένα θέμα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η διαφύλαξη του ευρώ είναι ε, επωφελής όχι μόνο για τα κράτη-μέλη, είναι προφανές αυτό και τα κράτη που δεν ε, συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ, αν το επιθεμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες για τη συγκρότηση του μονίμου μηχανισμού. Θα μπορέσουν επίσης ενδεχομένως να αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε δράσεις που θα βασιστούν στο μελλοντικό μηχανισμό, όπως έχουν ήδη κάνει κάποια κράτη ε, βάσει των προσωρινών ισχύοντων μηχανισμών. Προσπαθούμε να βρούμε μια σφαιρική απάντηση για την κρίση με τη συγκρότηση αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Ο ευρωπαϊκό μηχανισμό είναι ένα στοιχείο κλειδί και πρέπει να σημειώσουμε ταχύτατη πρόοδο. Αλλά θα σπεύσουμε βραδέω ε, και ε, προφανώς θα πρέπει να ε, προηγηθεί ένα συλλογικό προβληματισμός, να αντλήσουμε τα διδάγματα από την κρίση και να λάβουμε αποφάσεις καθοριστικής σημασίας για το κοινό μας μέλλον. Οφείλουμε να είμαστε σαφέστες σε σχέση με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Συμφωνούμε όλοι σχετικά με το ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε να διαφυλάξουμε τη γνωτοπιστωτική σταθερότητα, να αυξήσουμε την οικονομική σύγκληση των κρατών, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να επιτύχουμε την βιώσιμη ε, απασχόληση και ανάπτυξη. Ε, τώρα, αυτό το τρένο το αναπτυξιακό, ε, πάνω σε ποιες γραμμές θα κινηθεί, πάνω σε κοινοτικές γραμμές. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκή τροχιά για το αναπτυξιακό τρένο. Σπληρούνται ε, Σπληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να κάνουμε μία ε, απλουστευμένη μεταρρύθμιση ε, όπως προβλέπεται εξάλλου στο άρθρο 46 ε, της συνθήκης ε, αναρωτιούνται όλοι για το διακρατικό χαρακτήρα αυτού του μελλοντικού μηχανισμού. Κοιτάξτε, και εμεί θα προτιμούσαμε να προοδεύσουμε ταχύτερα και να βασιστούμε στο ισχύον σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ισχύουσα συνθήκη. Πλην όμω, λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν ε, ε, μειώνονται οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη νέα λύση θα έχουμε, αν θέλετε, βέλτιστε προποθέσει για να αντιμετωπίσουμε την κρίση για θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί ρητά μέσα στην ε, συνθήκη. Ε, θα ήθελα τώρα να τονίσω ω προ την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η γενική κατεύθυνση είναι μια πιο ενωμένη, μια ισχυρότερη Ευρώπη, αν θέλετε. Οπότε, βασικό στοιχείο είναι η αλληλεγγύη. Είναι μια θεμελιώδη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να είμαι σαφέστατο για αυτό το θέμα. Σε όλε τι συζητήσει που έγιναν για τροποποίηση τη συνθήκη, ε, υπενθύμεση επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επουδενή η τροποποίηση τη συνθήκη δεν μπορεί να ε, πλήττει το μηχανισμό αλληλεγγύη προβλέπεται στο άρθρο 122 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση ε, σοβαρών ε, προβλημάτων, σοβαρών απειλών που αντιμετωπίζει ένα κράτο μέλο. Ω εκ τούτου και αντίθετα με την άποψη που εκφέρουν διάφοροι, το άρθρο 120, 122 συγγνώμη, δεν τροποποιείται. Η ε, ε, αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως απόρρια την κοινή ευθύνη. Ε, είναι δύο αλληλένδετα στοιχεία ε, και μιλώντας για την οικονομική αλληλεγγύη και εξετάζοντας ε, τον προσωρινό μηχανισμό σταθερότητας, εξάλλου οι ίδιες διατάξεις θα ισχύσουν και για τον μελλοντικό μόνιμο μηχανισμό, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν τους ίδιους όρους ε, και να ακολουθούν μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχυθεί η προσπάθεια μέσω καλύτερου συντονισμού, καλύτερης εποπτείας. Αυτό ούτω ή άλλως είναι ένα από τα βασικά διδάγματα που αντλήσαμε από την κρίση. Στην ζώνη ευρώ, η πολιτική που θα ακολουθήσει η Ένωση θα αποτελέσει και το αίρισμα του μελλοντικού μηχανισμού ε, σταθεροποίηση. Οφείλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση του τέστην, να τη διευρύνουμε, να την εμβαθύνουμε για να κατοχυρώσουμε τη σταθερότητα τη ζώνη ευρώ, ε, ειδικότερα και γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό. Θα καλύπτονται όχι μόνο δημοσιονομικές πολιτικές αλλά και οικονομικές πολιτικές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εξάλλου αυτό είναι και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επί του οποίου έχουμε ήδη συμφωνήσει. Ε, δρομολογήθηκε η διαδικασία με την ε, υποβολή της έκθεση έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη. Φαίνεται σαφώς μέσα στο κειμένο ότι οι τωρινές πολιτικές δεν επαρκούν. Ε, θα πρέπει να καταβάλουμε ισχυρότερες προσπάθειες για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, να προσπαθήσουμε από κοινού να μην υπάρχει διάσταση δηλαδή να επιδιώκουμε μεγαλύτερη σύγκληση και να δημιουργήσουμε ε, νέα σημεία διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εξού και το πακέτο και οι έξι προτάσει που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τι οποίε γνωρίζω ότι θα ε, επιτύχουμε ε, την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού και τη διαδικασία προσπαθώντα να υλοποιήσουμε του φιλόδοξου ε, στα πλαίσια αυτών των μεταρρυθμίσεων εγγράφεται και αυτό ο μελλοντικό ε, μηχανισμό σταθερότητα, και σε αυτόν πρέπει να εγγραφεί και το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είμαι πεπισμένο ότι είναι ευέλτιστη προσέγγιση που προκρίνουμε και όλοι θα υπομισθούν τι δικέ του ευθύνε και το δικό του ρόλο και θα συμμετάσχουν δραστήρια στη συγκρότηση του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα. Δεν επαρκεί βεβαίω να έχουμε μια σωστή προσέγγιση. Πρέπει και να την εφαρμόσουμε ορθά. Σχετικά με την υλοποίηση λοιπόν και την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης, οφείλουμε να ακολουθήσουμε κάποιους ε, απλούς ε, κανόνες. Ε, Παραδείγματο χάρη ο κοινοβουλευτικός έλεγχος Επίση, ε, η νέα ισχύ που θα προκύψει από διαφανείς ε, νέου μηχανισμούς, νέα όργανα, ε, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια ω προς την οικονομική πολιτική της Ένωσης. Επίση, ισοτιμία, ισονομία αν θέλετε ενώπιον τη συνθήκης για όλα τα κράτη-μέλη. Είναι μια βασική αρχή. Οι δράσει που αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να πλήξουν την συνεργασία ε, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ολόκληρος ο σειρμός πρέπει να ακολουθήσει. Αν ξεφύγει εκτροχιαστεί ένα βαγόνι θα εκτροχιαστεί και ο σειρμός. Οφείλουμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα δηλαδή, στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μία ένωση και ως τέτοια θα πρέπει να δρούμε για να εξέλθουμε από την κρίση, να έχουμε ισχυρά θεμέλια για μία ανταγωνιστική, πιο ευημερούσα, σταθερότερη, αλληλέγγυα Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ε, θα αποφασίσουμε τις δράσεις μας. Ε, μέσα σε αυτό το πνεύμα ε, κινείται η Επιτροπή όταν πήρε τις αποφάσεις που πήρε και ανέλαβε τις δράσεις της και είμαι σίγουρος ότι θα τύχει τη υποστήριξή σας η πολιτική που εισηγούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντουρά Μπαρόζο. Τώρα, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε απολύτως καλά ότι χρειάζεται η ασφάλεια δικαίου να εξασφαλιστεί με βάση την τροποποίηση της συνθήκης. Χρειάζεται δηλαδή μια διαδικασία συνταγματικού χαρακτήρα για να εξασφαλίσουμε συνθήκες ασφάλειας δικαίου. Και γι' αυτό μιλούμε για την αναγκαιότητα τροποποίησης συνθήκης ώστε να εξασφαλιστεί και η σταθερότητα του ευρώ σε μόνιμη βάση. Και θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συστήσουμε άλλε δυνατότητε για περαιτέρω και διευρύτερε αναθεωρήσει τη συνθήκη και για την οικονομική πολιτική και μέσα στο ίδιο το άρθρο που θα μπορούσαν να γίνουν αναθεωρήσει ή τροποποίησεις διατάξεων ε, ή εδαφείων του ίδιου αυτού άρθρου με διαφορετικό πεδίο. Ωστόσο, ο κίνδυνο ε, μια τέτοια ευρύτερη αναθεώρηση θα ήταν να χρειαστεί να περάσουμε πάλι από τη διαδικασία των δημοψηφισμάτων και τι σχετικέ ε, δυσκολίε που θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη καθυστέρηση ακόμη ω προ την ε, διασφάλιση του ευρώ. Ωστόσο, η Δομισματική Ένωση είναι μια κοινότητα αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτήν την την κοινή αρμοδιότητα και ευθύνη να την διασπάσουμε μέσα από τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν πολλά, πολλά παραδείγματα όπου τα κράτη-μέλη μπορούν με ενισχυμένη συνεργασία να συμφωνήσουν σε νέους κανόνες και να ε, υποχρεώσουν τα θεσμικά όργανα να προβούν στα σχετικά μέτρα. Νομίζω ότι μπορούμε εδώ να ζητήσουμε μια δομή που να μην είναι μια παράλληλη δομή, γιατί θα ήταν εσφαλμένο να επιτρέψουμε την ανάπτυξη ε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, παράλληλων δομών γιατί αυτό θα αποτελούσε ένα κίνδυνο και διάσπασης και διχασμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει αυτή την εβδομάδα υπεύθυνα και με σοβαρότητα να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Μπορεί η κοινωτική μέθοδος να μην έχει την ίδια αξία. Η κοινοτική μέθοδος ε, Μάλλον η διακυβερνητική μέθοδος δεν μπορεί να εξισωθεί με την κοινοτική μέθοδο ως προς τις μεταρρυθμίσεις που μπορεί να φέρει. Αυτό το έχουμε δει και στο Σέγγεν και σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια βαθμιαία εξέλιξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την δυνατότητα για τα μέλη εκείνα, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ανήκουν ακόμη στο ευρώ, να γνωρίζουν ότι όταν έρθει η ώρα μπορούν σταδιακά να υπαχθούν σε αυτό το σύστημα και να έχουν την ίδια προστασία. Και το ίδιο σημαίνει μια σταδιακή προόδο προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας, της κοινή ανταγωνιστικότητας και της σύγκλησης. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τομέα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπου παραδοσιακά ισχύει η κοινοτική μέθοδος και η τροποποίηση της συνθήκης σημαίνει ταυτόχρονα ε, αποτροπή του κινδύνου της διάσπασης της ζώνης του ευρώ και εμείς ως Κοινοβούλιο αλλά και ως ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σοβαρή η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου ή της μεθεπόμενης Δευτέρας όπου οι καλούμεθα να δώσουμε το παρόν με ευθύνη και να καλέσουμε και το Συμβούλιο να δώσει το παρόν με ευθύνη. Εάν το Συμβούλιο λοιπόν δεχθεί μια διακυβερνητική λύση κατά τρόπο προσωρινό να ισχύσει, θα πρέπει να επιτρέψει ταυτόχρονα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσει το Συμβούλιο στην σχετική δράση και τις δράσεις που χρειάζονται. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίσουμε και μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μειωμένοι, κάποιοι βλέπουν ότι υφίστανται διακριτική μεταχείριση και ότι βρίσκονται σε μειονεκτούσα θέση, θα κινδυνεύουμε να τα ξαναδούμε μπροστά μας. Γι' αυτό θα πρέπει οι λύσεις να δοθούν εν εφέτο χρόνο και με πλήρη και διεξοδικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Εξω... Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολλές αδικαιολόγητες ε, καθυστερήσεις καθίσταται σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση που θα πρέπει να είναι αυστηρή για όσους δέχτηκαν το ευρώ. Εμείς ε, δεχόμαστε την ύπαρξη ενός ε, μηχανισμού σταθερότητας που θεωρούμε ότι είναι βασικό σκαλοπάτι για μία οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης, αν και έχουμε επιφυλάξεις πολιτικού και νομικού χαρακτήρα ως προς τη... τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Και χάρηκα διότι έμαθα ότι και εσείς συμμερίζεστε αυτές τις επιφυλάξεις. Αυτό όμως που μας απασχολεί είναι κάτι άλλο. Πώς θα δράσει ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα είναι ένα βήμα προς, τη, μια διακυβερνητική προσέγγιση που θα οδηγεί στη χρήση της διακριτικής ευχέρειας και ως προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του άξονα Γαλλίας-Γερμανίας θα πρέπει να δούμε πώς θα πλαισιωθεί και πώς θα οριστεί, δηλαδή πώς θα έχει ο μηχανισμός αυτός δυνάμει, θα κινηθεί δυνάμει του 136 που ορίζει ένα διακυβερνητικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να βασιστεί στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και η Επιτροπή θα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ μηχανισμού σταθερότητας και οικονομικής διακυβέρνησης. Επειδή όμως στην ε, διατύπωση του 136 δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ίχνος. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα ισχύσει ο μηχανισμός τώρα. Ποια διαδικασία θα ισχύσει για τη σταθερότητα του μηχανισμού, πώς θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ρήτρες αιρεσιμότητας, πώς θα συσταθεί η γραμματεία, τι γνώμη έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με αυτά που είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο ως προς το κύρος των έκτακτων μηχανισμών αλληλεγγύης θα διαδραματίσει ένα ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο μία επαναδιατύπωση του 136 ή μία δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί θετικά. Έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, ο κύριος Κίφερ Χόφστατ έχει το λόγο. Question, Mr. Gualtieri. Κύριε Γκουαλτιέρη, έχετε μία μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Γκουαλτιέρη, έχετε λάβει η υπόψη ότι η διακυβερνητική συνεργασία θα ήταν μία καλύτερη οδός για τους ανθρώπους, για τους πολίτες Ευρώπης και ιδιαίτερα τους ε, άνεργους σε σχέση με ένα υπερκράτος υπέρ του οποίου τάσεστε. Αυτό το σκεφτήκατε ποτέ, Γκουαλτιέρη. Ε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται από τις συνθήκες και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ε, ρόλος μας να ανταποκριθούμε ως, ως άμεση εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Φερχόφστατ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μπαρόσο για την ε, τροποποίηση της συνθήκης. Ε, προφανέστατα τώρα θα αποφανθούμε κι εμείς ε, και ελπίζω πριν την 24η Μαρτίου γιατί είναι πολύ, σημαντική, πολύ σημαντικό το Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα τότε. Απλουστευμένη διαδικασία. Αυτή θα επιλέξουμε. Θα δούμε. Ε, πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι. Ο πρώτος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι προσπαθούμε να επιτύχουμε το εξή. Ο μηχανισμός αυτός ε, να, αποτελεί, να ε, τον διαχειρίζεται μάλλον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδατε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο εξέδωσε 5 δις ευρωμολόγων στις 6 Ιανουαρίου. Και το ίδιο έγινε σε διακυβερνητικό επίπεδο στις 25 Ιανουαρίου, 5 δι σε πενταετή ευρωομόλογα. Το ίδιο ακριβώς. Τα ευρωομόλογα της ε, ε, Επιτροπής ήταν με 2,5% ενώ το διακυβερνητικό σύστημα εξέδωσε ομόλογα 2,89%. Άρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, που διαχειρίζεται η ενωσιακή μέθοδος επιτυγχάνει χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με το διακυβερνητικό σύστημα. Ήθελα να το υπενθυμίσω, είναι σημαντικό. Η μέθοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όπως προκύπτει σε σχέση με το διακυβερνητικό σύστημα. Δεύτερον, ε, οφείλουμε να αναρωτηθούμε ε, αν μπορούμε να τροποποιήσουμε το άρθρο 136 ούτως ώστε να ενισχύσουμε το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης ε, που ε, είναι επιτάπητος. Η κυρία Κόλ και οι συζητητές έχουν υποβάλει έξι προτάσεις αλλά πέρα από αυτές τις έξι προτάσεις θέλουμε και το πράσινο φως από το Συμβούλιο για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα με το άρθρο 136. Δηλαδή να πούμε ότι αν ε, ε, χρησιμοποιήσουμε το μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπιση κρίσεων, δηλαδή το άρθρο 136, τότε αυτόματα μπορεί να δρομολογήσει τη διαδικασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι εφικτό ε, να υπάρξει ανασταλτική μειοψηφία, αν θέλετε, στο Συμβούλιο και να μπλοκάρει τη διαδικασία. Δεύτερη παρατήρηση που μάλλον θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότησή μα και στρέμουμε προ τον κύριο Μπρό και τον κύριο Γουαλτιέρη που είναι συνεισηγητέ για την Επιτροπή μα. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Ε, Κύριοι Μπρόκ και Γουαλτέρη, με την ιδιότητα των εισηγητών, θα πρέπει να προσπαθήσετε να ε, ε, έχετε κάποιε διαβεβαιώσει του Συμβουλίου, κάποια εχέγγυα, γιατί το τωρινό πακέτο, κυρίω αυτά που εξήγηλαν τι τελευταίε ημέρε, σύμφωνα ανταγωνιστικότητα, διακυβερνητική μέθοδο, πολλές χώρες ε, καταψηφίζουν ε, την πρόταση. Υπάρχει πραγματική διχογνωμία, διάσταση απόψεων στο Συμβούλιο και νομίζω ε, ότι χρειαζόμαστε κάποιες διαβεβαιώσεις από το Συμβούλιο. Σε αυτό το δεύτερο πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης θα συμπεριλάβουν και την μέθοδο της Ένωσης. Γιατί? Διότι η διακυβερνητική δεν λειτουργεί. Για φανταστείτε, παραδείγματο χάρη, αν οι κανόνε περί ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο αντικείμενο διαχείρισης ε, του Συμβουλίου. Θυμηθείτε πόσε φορέ έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσει επειδή δεν τηρούνται οι κανόνε ανταγωνισμού. Ε, λοιπόν, αν το αναλάβει το Συμβούλιο, ποτέ, ποτέ, σα διαβεβαιώ, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο σε επιχείρηση επειδή δεν τηρεί του ε, κανόνε ανταγωνισμού. Και το ίδιο ισχύει και για το μηχανισμό κρίση ε, και γι' αυτό σα λέω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εχέγγυα από το Συμβούλιο ότι μέσα στο δεύτερο πακέτο οικονομική διακυβέρνηση θα υπάρχει η μέθοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, κύριε από τους Πρασίνους τώρα η συμπρόεδρος κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, είναι σαφές νομίζω ότι το Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους προχωρεί με την απλουστευμένη διαδικασία τώρα αυτή η αναθεώρηση της συνθήκης. Είναι σαφή οι λόγοι και πιεστικοί οι λόγοι. Ταυτόχρονα όμως είναι και σαφές το ότι το Κοινοβούλιο δεν θεωρεί σωστή την επιλογή μιας μεθόδου με την θέση εφαρμογή του μηχανισμού κρίσης που θα μπορούσε ενδεχομένω να οδηγήσει στο μέλλον την, ε, στη λήξη της ε, κοινοτικής μεθόδου και θα άφηνε πεδίο ε, δράσει αποκλειστικά και μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό έχουμε επικριτική στάση έναντι της ε, διαφαινόμενη ενίσχυσης της διακυβερνητικής μεθόδου. Θεωρούμε ότι στην Ευρώπη οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, καταλαβαίνουν όλο και λιγότερο τι συμβαίνει, τι αποφασίζεται, υπό ποιους όρους. Οι Γερμανοί στρέφονται κατά τον Ελλήνων. Οι Έλληνες στρέφονται κατά των Γερμανών, εξοργίζονται, ε, οι μεν κατά των τραπεζών, οι δε κατά των επιχειρήσεων. Δεν οφείλεται αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στην διακυβερνητική, στο μαύρο αυτό κουτί που ονομάζεται Συμβούλιο όταν λαμβάνουν αποφάσει. Με περισσότερη μόνο διαφάνεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, αλλιώ θα χάνουμε όλο και περισσότερο το έδαφος της αξιοπιστίας μας, το έδαφος της εμπιστοσύνης των πολιτών. Θα το χάνουμε κάτω από τα πόδια μας με ραχδαίους ρυθμούς. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ μας προτείνετε εσείς βέβαια την απλουστευμένη αυτή μέθοδο, αλλά θα σα παρακαλούσα να μην λησμονήσετε ότι θα πρέπει να περιοριστεί αυτή στο ελάχιστο. Το ΔΕ Συμβούλιο και η Επιτροπή να μην λησμονήσουν πως εκπρόσωπος των πολιτών είναι το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο και θα πρέπει η εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας και η όποια ε, αναθεώρηση, μικρή μεταρρύθμιση να γίνει με βάση τα όσα έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες Ευρώπης. Δηλαδή περισσότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το μέλημά μας. Εάν δούμε τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα, όπου γίνεται λόγος ακόμη και για ιδιωτικοποίηση των ακτών των παραλίων προκειμένου να αποπληρωθεί το χρέος, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν ακραίες απόψεις, μια λιτότητα ακραία που επιβάλλεται από την Γερμανία και που οδηγεί τα κράτη αυτά που έχουν υψηλό δημόσιο έλλειμμα στο χείλος της καταστροφής. Αυτά πρέπει εξάπαντος να αναθεωρηθούν το ταχύτερο δυνατό και η κρίση να αντιμετωπιστεί με πραγματικά και ουσιαστικά αλληλέγγυες πολιτικές. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Μόνο έτσι μπορεί η Ευρώπη να αντιληφθεί τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη μεγάλη κρίση. Και ακόμη θα ήθελα να συμπληρώσω ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε στην επίδειξη και ένδειξη αλληλεγγύης προς άλλα ακόμη κράτη της Ευρώπης, γιατί το ταμείο που έχουμε τώρα στη θέση μας δεν θα επαρκέσει. Έχει αποφασιστεί περισσότερη ρευστότητα να εξασφαλιστεί στο πεδίο αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και για τα ευρωομόλογα θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε να συζητήσουμε. Ο κύριο ε, Φερχόφστατ ήδη έδωσε μια σαφέστατη αιτιολόγηση και βάση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Όχι, θα πρέπει να συζητήσουμε το μέλλον μα και την ισοδηματική μα πολιτική από εδώ και εμπρό. Και ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ, πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερο χώρο για συζήτηση, έτσι ώστε εν τέλει να την διεξαγάγουμε σε κάθε τη διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εκ μέρους των μεταρρυθμιστών ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω τις αλλαγές της συνθήκης και θα υποστηρίξει τις αλλαγές και η ομάδα μου, διότι θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέλος του ευρώ και ελπίζω ποτέ να μην προσχωρήσουμε. Το ίμιση του εμπορίου μας αφορά ε, συναλλαγές με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Το City του Λονδίνου είναι η καρδιά των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ελπίζουμε ότι αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας θα, θα μας υποστηρίξει μέσω και μακροπρόθεσμα. Ελπίζουμε λοιπόν να δράσουμε υπεύθυνα και να εγκρίνουμε την αλλαγή που πρότεινε το Συμβούλιο. Αλλά εάν το ευρώ επιμερίσει στο μέλλον, θα πρέπει να γίνουν πιο καινοτόμε αλλαγέ. Κύριε Μπαρόζο, μπορείτε να κάνετε όποια εποπτεία θέλετε, η οικονομική διακυβέρνηση. Αλλά επί τη ουσία, εάν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία παραμείνουν μέσα στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να γίνουν τόσο ανταγωνιστικές όσο και η Γερμανία. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ. Επόμενο μιλητή είναι ο κύριο Λόταρ και από την Αριστερά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει μικρό διάστημα ζωή, πλην όμω τώρα και μέσα σε μερικού μήνε από τη θέση εφαρμογή τη, ε, καλούμαστε να την τροποποιήσουμε για δεύτερη φορά και μάλιστα με ισχυρισμούς κατεπίγουσες ανάγκες που σημαίνουν ότι δεν μπορεί να ε, υπαχθεί στους συνήθεις ε, δημοκρατικούς κανόνες για την τροποποίηση. Πρέπει με ταχεία διαδικασία δηλαδή να αναθεωρηθεί. Είδαμε πως ε, η ομπρέλα διάσωσης, το δίκτυ διάσωσης των δισεκατομμυρίων ευρώ για τις τράπεζες πέρασε μέσα από ταχείες διαδικασίες κατεπίγοντας το Κοινοβούλιο. Τώρα το Συμβούλιο ασκεί και πάλι πιέσεις χρονικές και ορισμένες κυβερνήσεις θέλουν από ό,τι φαίνεται να ε, προχωρήσουν σε μια ταχύτατη αναθεώρηση συνθήκης. Η ομάδα μας απορρίπτει τέτοιου είδους ε, δράσεις πιεστικά χρονοδιαγράμματα και απαιτεί τροποποιήσεις της Λισαβόνας να γίνονται μόνο με βάση τα όσα προκύπτουν από τις συνήθεις διατάξεις αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, εκ μέρου της Ευρώπη των Ελευθεριών και Δημοκρατιών ο κύριος Earl of Dartmouth. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε ως τελωνιακή ένωση. Απλά πράγματα. Στη συνέχεια έγινε πολιτική ένωση, αλλά δεν υπήρχε ε, η συγκατάθεση του λαού. Δεν ήταν δημοκρατική. Κατόπιν έγινε νομισματική ένωση. Ε, τέλος πάντων, ένωση. Δέκα μήνα απ' έξω, γιατί ήταν λογική. Τώρα τι έχουμε, μια ένωση χρεών. Ε, μια ένωση χρεών, μια χρεωμένη ένωση που δεν λειτουργεί. Για να δούμε τώρα το επιτόκιο ε, της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας. Αν λειτουργούσε εύρυθμα η, Νομισματική Ένωση, όλα τα μέλη τη Ένωση, όλε οι χώρε στη ζώνη ευρώ θα μπορούσαν να δανείζονται με το ίδιο ε, επιτόκιο όπω το βασικό, δηλαδή το κεντρικό επιτόκιο τη ε, ε, Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν συμβαίνει όμω αυτό. Η Πορτογαλία πληρώνει 4,28% περισσότερο από τη Γερμανία. Η Ιρλανδία 5,9% περισσότερο από τη Γερμανία. Η Γαλλία 8,25% περισσότερο από τη Γερμανία. Ε, είναι και βρισκόμαστε μια καμπή. Δεν ε, περιμένω από τον πρόεδρο του ΕΛΚΕ ή από τον πρόεδρο των Σοσιαλιστών να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα αλλά πιστεύω ότι λίγαν συντόμω θα αναγκαστούν να καταλάβουν το πρόβλημα σα, ε, γιατί δικό σα είναι το πρόβλημα κυρίω, ε, θα λυθεί καλύτερα μέσω διακυβερνητικής ε, συνεργασίας. η οικονομική διακυβέρνηση είναι μια παγίδα. Αφήστε που δεν έχετε καμία εντολή. Κανεί δεν αναφέρθηκε ή εν πάση περιπτώσει το καν το σκέφτηκε κατά πώ φαίνεται ότι πιέζονται σκληρά οι φορολογομονοί όλων των κρατών μελών ενώ εσείς επιχειρείτε και ματαιοποιείτε προσπαθούν να οικοδομήσετε αυτή την οικονομική αυτοκρατορία. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν 27 κράτη-μέλη και 11 από αυτά ε, σαφέστατα συνεισφέρουν στον ε, προπολογισμό της Ένωσης ε, και οι υπόλοιποι απλώς ε, είναι αποδέκτες των χρημάτων. Υπάρχουν αυτοί που συμμετέχουν ε, και αυτοί που δεν συμμετέχουν λοιπόν, ο Γερμανός φορολογούμενος, είμαι σίγουρος ε, ότι δεν θα ανέξει για πολύ περισσότερο για αυτή την κομμωδία, την οικονομική κομμωδία. Ο William Jennings Bryan το 1896 είπε σε μια διάμεση ομιλία του «Δεν θα σταυρώσετε την ανθρωπότητα πάνω σε ένα χρυσό σταυρό». Σήμερα λοιπόν σας λέω εγώ ε, και απευθύνομαι κυρίως στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν, ε, λέω λοιπόν, δεν θα σταυρώσετε ε, τους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Λυπής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σταυρό του ενίου νομίσματος. The next speaker, Mr. Bruno Ευχαριστώ πολύ, μιλήσω, ο κύριος Bruno Γκολνής. Καταρχάς, για το σκάνδαλο της λεγόμενης απροστευμένη διαδικασίας. Ουσιαστικά, μια εγκρυπτό και παραβίστο τροποποίηση των συνθήκων, χωρί ανοιχτή διαβούλευση και ε, διαβούλευση με του πολίτε Ευρώπη. Και όμω έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί πρόκειται για την ε, διαιώνιση του σταθεροποιητικού ταμείου και τη δημιουργία ενός ε, κοινού χρέους από κράτη ήδη υπερχρεωμένα τα οποία δεσμεύονται να αποπληρώσουν αυτό το χρέος πριν έχουν αποπληρώσει το εθνικό τους ε, χρέος είναι σαν την περίφημη υπόθεση του λεγόμενου πυροτεχνουργού Καμαμπέρ, ενό ε, ήρωα ε, κινούμενων σχεδίων στη Γαλλία, ο οποίο πήγαινε να κλείσει μια τρύπα μέσα στο στρατόνα που και για να την κλείσει έσκαβε, έσκαβε, έσκαβε και έπαιρνε χώμα από δίπλα του και έτσι άνοιγε μια άλλη ε, τρύπα δίπλα. Εδώ λοιπόν η ανταγωνιστικότητα και βλέπουμε και από το Γενικό Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Γενικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γαλλικού κράτους ένα μνημόνιο το οποίο δείχνει ότι τα μέτρα δεν θα είναι καθόλου ανώδυνα, θα είναι υψηλή επιβάρυνση εποπτεία, σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λιτότητα, σύγκληση σε όλες τις πολιτικές και παραθέτω εδώ που έχουν επίδραση στην ανταγωνιστικότητα ακόμη και να έχουν να κάνουν με τομείς εθνικής αρμοδιότητας αποκλειστικά. Δηλαδή σε όλη τη ζώνη ζώνη ευρώ θα επιβληθούν οι γερμανικές πολιτικές που προσφέρουν οράματα και όνειρα στον κύριο Σαρκοζή. Δηλαδή θα διαιωνιστεί το εθνικό χρέος μέσα από τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό και θα δημιουργηθεί ένας ειδικό φόρος για να το χρηματοδοτήσει. Το, το, έχουμε πάρει τελείω λάθος δρόμο, Άλλος, άλλα πράγματα θα πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος Μπαρόσο έχει το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις. Merci les rapporteurs, et θα ήθελα να συγχαρώ τους συζητητές Μπροκ και Γκουαλτιέρη και θα ήθελα να τους επισύρω την προσοχή σε μια ενδεχόμενη διακυβερνητική ολίσθηση. Ας είμαστε σαφείς. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή υποστήριξε αυτή την αναθεώρηση διότι πιστεύουμε ότι πράγματι πρόκειται για ένα τρόπο για να ανταποκριθούμε σε μία πρόκληση μέσα στα πλαίσια μιας αρμοδιότητας η οποία δεν προβλεπόταν από τη συνθήκη, δηλαδή η συνθήκη δεν προέβλεπε ένα μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας. Γι' αυτό έπρεπε ομόφωνα να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό σε διακυβερνητική βάση. Επρόκειτο για ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών και δεν σας κρύβω και το λέω σαφώς ότι θέλω να πάμε πιο γρήγορα. Γιατί ένα βήμα καθαρά διακυβερνητικού χαρακτήρα είναι πρόοδος, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι κάναμε πολλά βήματα με βάση αρχικά τη διακυβερνητική, όπως για παράδειγμα το Σέγγεν ή τον χώρο δικαιοσύνης και ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να βασιστούμε σε κάτι το οποίο δεν βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο καθαρά, αλλά αποτελεί ενίσχυση της συλλογικής δυνατότητας να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις οι οποίες δεν προβλέπονταν από τη συνθήκη και η απάντησή μας είναι θετική. Θα πρέπει να απαντήσουμε καταφατικά. Γι' αυτό η άποψη της Επιτροπής είναι θετική σε σχέση με αυτή τη μεταρρύθμιση της συνθήκης, αλλά η Επιτροπή προτιμά την κοινοτική προσέγγιση. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε και κατά την προπαρασκευή αυτής της απόφασης. Πολλοί είχαν προτείνει να αλλάξουμε το άρθρο 122, δηλαδή να απολύψουμε μία αρμοδιότητα που προβλεπόταν από τη συνθήκη της Ρώμης. Εγώ αντιτάχθηκα τότε και μπορώ να πω ότι αυτή η νέα αρμοδιότητα την οποία τώρα μπορούμε να αναπτύξουμε μπορεί στρίκτο σένσου να μην αφορά την κοινοτική μέθοδο αλλά ενισχύει τις εξουσίες μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, νομοθετικές ή έτσι ώστε να εγγυηθεί αυτό τον μηχανισμό στα πλαίσια της Ευρωζώνης με βάση τις αρμοδιότητες και εξουσίες που απορρέουν από τις συνθήκες. Αυτή είναι μια απόλυτα σαφής θέση. Ορισμένοι στη συζήτηση, κατά τη συζήτηση μίλησαν για διαφορές μεταξύ των κρατών μελών δηλαδή μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωζώνης. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες διαφορές και η βασική είναι ότι στην Ευρωζώνη το χρέος είναι χαμηλότερο από το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υψηλότερο από το χρέος της Ευρωζώνης. Αλλά εδώ μιλάμε και για θέμα σχετικής ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό αποζητούμε μία λύση για τη σύγκληση της ανταγωνιστικότητας και εάν και μερικοί δεν συμφωνούν, αφήστε μας να κινηθούμε προς μία σύγκληση της Ευρωζώνης για αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν. Διότι δεν μιλάμε μόνο για τους φεντεραλιστές οι οποίοι θέλουν περισσότερη διακυβέρνηση. Το ζητάν και οι ίδιες οι αγορές, ζητάν αυτή την οικονομική διακυβέρνηση. Σήμερα οι αγορές ζητούν όχι μόνο την αποφασιστικότητα στην υπεράμυνα του ευρώ, αλλά και έναν τέτοιο μηχανισμό. Διότι δεν αφήνουμε τις τύχες μας στα χέρια των dealer. Γι' αυτό χτίζουμε άλλα θεμέλια με βάση την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα, αλλά αυτή θα είναι μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε μια άλλη μέρα. Η Επιτροπή έχει αποφανθεί καταφατικά για αυτή τη μεταρρύθμιση της συνθήκης, ζητώντας από τους πάντες να μην δημιουργήσουμε ε, μηχανισμούς που όπως είπε ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ρήξεις ή διχασμούς. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την ένωση καθεαυτή, την ύπαρξή της, γιατί εμείς ε, δρούμε και υπέρ της Ευρωζώνης αλλά και υπέρ των άλλων που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Άρα για να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις ας μην δημιουργήσουμε προηγούμενα που θα δημιουργήσουν μελλοντικές ε, ρήξεις. Ας εγγυηθούμε το, την Ένωση, την ίδια την ύπαρξη της Ένωσης μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητα. Σας ευχαριστώ. Ε, από τους άλλους ομιλητές, ο κύριος Μάνφρετ Βέμπερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απαραίτητη και ορθή τροποποίηση τη συνθήκη και η θεσμική συζήτηση που διεξάγουμε αποδεικνύουν ότι μέσα σε ένα χρόνο η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, δεν είναι πλέον σε θέση να επιλύσει τι μεγάλε προκλήσει που παρουσιάζει ο κόσμο στη σύγχρονη εποχή. Αυτό αποδεικνύει αυτή η συζήτηση και ταυτόχρονα βλέποντα τη συνθήκη την οποία συζητούμε σήμερα, ε, διαπιστώνουμε ότι η Βρετανία, Τσεχία, προχωρούν σε συζητήσεις ευρύτατο δημόσιο διάλογο για τη συνθήκη που θα ήταν πριν αδιανόητε. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με πεδία τάσεω πολύ σημαντικά με οποία κινούμεθα, μέσα από τα οποία πρέπει να ξεφύγουμε γιατί διαφορετικά δεν μπορεί το εθνικό κράτο να δώσει απαντήσει. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να μιλήσει και ο πολίτη αντιλαμβάνεται ότι είναι μεγάλε οι προκλήσει και ότι από την Ευρώπη θα δοθούν αυτέ οι απαντήσει. Έτσι μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι μεγάλε προκλήσει, και γι' αυτό χρειάζεται να είναι ισχυρή η Ευρώπη. Και υπάρχει ένα ακόμη πιο σημαντικό ερώτημα, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τι φέρει εν τέλει προς τα μπρος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το όραμα της Ευρώπης, τι είναι αυτό που το κάνει να ζει και να ανδρώνεται. Είναι η, η ειρήνη, είναι το όραμα και η βεβαιότητα της ειρήνης όλα αυτά τα χρόνια και τις δεκαετίες που έχουμε ζήσει μαζί. Η βεβαιότητα ότι δεν θα ξαναπέσουμε στον πόλεμο. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να προβάλλουμε ακριβώς αυτό το επιχείρημα, η παγκοσμιοποίηση με τα αρνητικά επιχειρήματα με τα οποία μερικές φορές ε, περιγράφεται. Ίσως θα μπορούσαμε να πείσουμε τον πολίτη, να αγγίξουμε την ψυχή του μιλώντας του τι για το τι σημαίνει ευρωπαϊκό όραμα, τι καθήκον έχει αναλάβει η Ευρώπη αυτή η κοινή. Οι Ευρωπαίοι οι Βραζιλιάνοι, οι Αμερικανοί, οι Ιάπωνες θέλουν τώρα να είναι σε θέση να ζήσουν μαζί. Και εμείς σηκώνουμε το χέρι σε αυτόν τον κοσμιοποιημένο κόσμο και λέμε έχουμε λάβει υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί οι Κινές δεν πρέπει να συστήσουν αυτά. Ή σηκώνουμε το χέρι και λέμε έχουμε λάβει υπόψη τα μελήματα για το περιβάλλον, γιατί δεν πρόκειται να συστήσουν οι Αμερικανοί. Ε, έχουμε λάβει υπόψη τα ζητήματα και την ε, ανέμακτη ε, και ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτά όλα μπορεί να τα προσφέρει η Ευρώπη. Κοιτώντα με μια ματιά προ την Τινησία, καταλαβαίνουμε τι είδου πρότυπο μπορούμε να αποτελέσουμε. Βλέπουμε κράτη τα οποία αγωνιούν να μοιάσουν σε εμά, στα δικά μα κράτη. Είμαστε υπόδειγμα για του άλλου. Και γι' αυτό νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε για το όραμα, για, το, για την ευρύτερη εικόνα, για το μεγάλο πίνακα που σημαίνει όχι εθνική ε, αποδοχή αλλά πανευρωπαϊκή και παγκόσμια αποδοχή. Ευχαριστώ. Κύριε Βέμπερ, συμφωνείτε να σα τεθεί ένα ερώτημα με τη διαδικασία του δελτίου, Κύριε Ντερόσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Ντερός, κύριε Βέμπερ, ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτησή μου. Ελπίζω δε ότι επί τη ευκαιρία θα την απαντήσει και ο κύριος Μπαρόσο, ο πρόεδρο Μπαρόσο, γιατί ουσιαστικά σε αυτόν απευθύνεται. Η ε, τροποποίηση αυτή τη συνθήκη βεβαίω μα απασχολεί ω προ τη διαδικασία τη. Αυτή η απλουστευμένη διαδικασία δίνει τη δυνατότητα και στα 27 εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα τουλάχιστον τη σύμφωνη γνώμη στην έγκριση αυτή τη ε, τροποποίηση. Και προβλέπεται ένα εξάμεινο για τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να λάβουν τη σχετική απόφαση. Εσείς λέτε ότι πρέπει η απόφαση να υιοθετηθεί, απόφαση του Συμβουλίου, που ελήφθη τον Δεκέμβριο πρέπει να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Πώς θα γίνει αυτό, τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο κύριος Βέμπερ. Ε, πολύ ευχαριστώ να απαντήσω. Έχετε δίκαιο ότι τα κράτη-μέλη είναι η κυρίαρχη των συνθήκων. Εκείνα λοιπόν καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την τροποποίηση και επίσης σε πολλά από τα αισθήματα τα οποία εγώ προσπαθώ να θίξω βλέπουμε πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε σε όλη αυτή τη δικασία αρκετό χρονικό περιθώριο ώστε να οριμάσει και να προχωρήσει και να δώσει και στους πολίτες απαντήσεις στις αγωνιώδεις ερωτήσεις που τους απασχολούν. Δεν βλέπω πρόβλημα λοιπόν ως προς το ζήτημα του χρόνου. Πρέπει να δώσουμε σωστές απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος κύριο Σούλτς είναι ο επόμενος. Έχω λάβει μια επιστολή ε, εκ μέρους σας κύριε Πρόεδρε, κύριε Σούλτς εάν υπάρχει κάποια παρεξήγηση ως προς τον κατάλογο, ως προς τη σειρά δηλαδή των ονομάτων στον κατάλογό μας, ευχαριστώ να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ο κύριο Σούλτ. ναι πρόεδρε ήταν προσωπική επιστολή προς εμά και όχι προς το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ όμως που μου δίνετε το λόγο έστω και με καθυστέρηση. Ίσως θα μπορούσαμε και στα εσωτερικά μα, στον εσωτερικό μα κανονισμό δηλαδή, να, να προχωρήσουμε σε ορισμένε τροποποίησεις επί τη ευκαιρία αυτών των τροποποίησεων στη συνθήκη. Εν πάση περιπτώσει, τροποποίηση συνθήκη λοιπόν είναι περίπλοκη... έστω και η απλουστευμένη διαδικασία για τροποποίηση συνθήκη, είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Και αυτό ε, μας δείχνει πόσο, σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε, περίπλοκη κατάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση ακόμη και η απλουστευμένη διαδικασία να αποτύχει. Να αποτύχει, να καταρρεύσει δηλαδή Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα περιπέσουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει να διαρωτηθούμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να μην αποτύχει αυτή η αποστευμένη διαδικασία. Και το άλλο ερώτημα που έχει να κάνει με τη διάσωση όχι αυτή τη αποστευμένη διαδικασία αλλά ολόκληρου του ευρωπαϊκού εγχειρήματο βρίσκει την απάντησή του σε μια συλλογική και συνεκτική στάση και δράση από πλευρά όλων μα. Και γι' αυτό θα ήθελα να προσθέσω τρει βασικέ σκέψει, βασικέ και ουσιώδει κατά την άποψή μου. Ύστερα από την έναρξη αυτή τη σοβαρότατη κρίση, ερωτώ ποια είναι η εξωτερική αξία του νομίσματός μας, του κοινού μας νομίσματος. 1 δολάριο και 35 ευρώ. Ένα και 17 δολάρια ήταν η αξία του όταν εισήχθη. Τώρα είναι στα 1,35. Βλέπουμε την αξία ενός νομίσματος όταν είναι ισχυρό, όταν είναι διεθνές νόμισμα βλέπουμε την αξία του να διατηρείται και να ενισχύεται. Εδώ και ένα χρόνο το, ευρώ είναι γερό νόμισμα, είναι σταθερό νόμισμα και ο μόνος λόγος αποσταθεροποίησής του είναι η διπλοκλωσία των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις οι οποίες κρύβουν το κεφάλι στην άμμο και δεν το στηρίζουν. Τα μέσα υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια κοινή μέθοδο δράσης. Και όταν πούμε όταν λέμε Ευρώπη, μην μου πείτε, όχι εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε εμεί, δεν είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κυβερνήσει, τα ε, κυρίαρχα κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει προς τα έξω ζώνες νομισματικές ισχυρές, γέρες, που όμως δεν είναι σε θέση προς τα έσω να διαφυλάξουν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα νόμισμα γερό, μια νομισματική πολιτική ισχυρή με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια ταυτόχρονα. Και η δεύτερη παρατήρηση. Αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ευρώπη συμβαίνουν στο πλαίσιο των συνθήκων. Μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων λοιπόν και όχι έξω από αυτό, όχι αυθαίρετα. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι μέσα από τις συνθήκες, μέσα από το πλέγμα των συνθήκων, τότε για μας τους πολίτες κεντρική σημασίας θα πρέπει να είναι ο ρόλος εκείνου του οργάνου που έχει το ρόλο του θεματοφύλακα των συνθήκων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομιμοποίηση για δράση έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αναφορά φυσικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάμει των συνθήκων. Και πολύ σωστά αναφέρατε εσείς αυτά που αναφέρατε όπως και ο κύριος Μπρόκος και ο κύριος Γουαλτιέρη. Και επίσης, τρίτη παρατήρηση, κίνδυνος για την Ευρώπη είναι το να είμαστε ο ισχυρότερος οικονομικός χώρος της, ε, του κόσμου με 500 εκατομμύρια πολίτες και να μην δρούμε ενωμένα αλλά να αναλαμβάνουμε δράση και αποφάσεις σε 27 χωριστά κομμάτια που στρέφονται το ένα κατά του άλλου, στρέφει το ένα την πλάτη στο άλλο. Αυτό το βλέπουμε και στην νότια όχθη της Μεσογείου. Βλέπουμε ότι προσπαθούν όλοι να μοιάσουν σε εμάς. Η Ευρώπη είναι ο κοινωνικός κινητήρας, το πρότυπο το κοινωνικό για όλο τον κόσμο και θα πρέπει να συζητήσουμε αν θέλουμε αυτή η Ευρώπη να έχει μέλλον ή αν θα παραπέσει στην εθνική κυριαρχία, τις εθνικές αρμοδιότητες και τον κατακαιρματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ιβο Στρέιτσικ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Όποιες και να είναι οι σχέσεις μας με το κοινό νόμισμα, το ευρώ, νομίζω ότι όποιος ε, ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την στερότητα της Ευρωζώνης. Χρησιμοποιούμε αυτό το νόμισμα διότι οι οικονομίες μας είναι αλληλένδετες. Και όταν ο πρόεδρος Μπαρόζο μίλησε για τον μηχανισμό σταθερότητας, μίλησε για καλύτερη εποπτεία για οικονομικό συντονισμό, για συντονισμό φορολογικών πολιτικών και για συντονισμό κοινωνικών πολιτικών. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε το δρόμο για μια φορολογική ένωση και ποτέ δεν ζήσαμε μια τέτοια ένωση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ανακύψει μια φορολογική ένωση θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική. Άρα μπορεί να μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι από πολιτικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει μία μετάλλαξη. Ρωτήστε τους Ευρωπαίους πολίτες τι θέλουν, γιατί εδώ και δεκαετίες δέχονται παθητικά και δεν αποφασίζουν. Ο κύριος Higgins, ένας νέος μηχανισμός σταθερότητας προτείνεται στην προεκλογική εκστρατεία στην Ιρλανδία. Αυτή που θα απαρτήσουν τη νέα κυβέρνηση μιλάνε για νέα μέτρα μέσα στα πλαίσια και τη συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά αυτό δεν αποτελεί παρά εικασίες και δεν θα πρέπει οι Ιρλανδοί να ψηφίσουν για ένα νεφέλωμα εικασιών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαρόσο και να του πω το εξής, να μην παρέμβει στην προεκλογική αλλά να δίνει πραγματικές πληροφορίες στον ε, ε, Ιρλανδικό λαό. Ο ε, ο Επίτροπος Ρεν είπε ότι μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά αυτό αφορά μια νέα κυβέρνηση και πριν μπει σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός του 2013 και αυτό σημαίνει μείωση των επιτοκίων. Επίσης, οι κερδοσκόποι θα αναλάβουν τα, τις ζημίες τους και δεν θα σταυρώσουν τον ε, Ιρλανδικό λαό. Επίσης, μέσα στα πλαίσια των επενδύσεων θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, διότι διαφορετικά θα κατασπαραχθεί η κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Νικόλ Σίνκλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάλι τα ίδια. Το ευρώ μας οδήγησε στη διπλή μεταρρύθμιση της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνθήκη αθέτησε το δημοψήφισμα της ε, ε, Ιρλανδίας και βεβαίως τη δεύτερη φορά μας δόθηκαν λάθος πληροφορίες για να ψηφίσουμε. Και τώρα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, η Ευρώπη δεν κάνει ένα βήμα πίσω για να δει πού έσφαλε. Θέλετε τα μικρά κράτη να πληγούν περισσότερο. Θέλετε να τα προσδέσετε σε αυτό το άρμα με μεγαλύτερες δυσκολίες μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει ένα θέμα χρέους, αλλά δεν πρέπει, ε, δεν πρέπει παρά να διασώσει άλλες χώρες, όπως την Ιρλανδία, ιδιαίτερα όταν ε, πρέπει να δανειστούμε αυτά τα χρήματα. Η κυρία Κέι Σουίνμπερν έχει το λόγο. Το να αλλάξουμε τη συνθήκη δεν είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ελαφρά την καρδία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θα τροποποιήσουμε τη συνθήκη. Η συνθήκη πρέπει να αλλάξει για να προστατευτούν οι χώρες της Ευρωζώνης. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η θέση αυτών που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, έτσι ώστε με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να αντιμετωπίσουμε και τα μεγάλα ελλείμματα ή το υψηλό χρέος, το οποίο δεν θα μειωθεί. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο έτσι ώστε η Ευρωζώνη να μπει σε μία τάξη αυτό αφορά και τις άλλες χώρες. Η κάθε χώρα θα πρέπει να δει τη φορολογική του, της πολιτική και να ενισχύσει την οικονομία της. Και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την πραγματική μεταρρύθμιση. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική ανταγωνιστικότητας. Ο κύριος Σεύκοβης έχει το λόγο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, υποστήριξη που προσέφεραν σχετικά με τη μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα εξασφαλίσει μια ισχυρότερη Ευρώπη και θα κατοχυρώσει τον μελλοντικό μηχανισμό που είναι και το αντικείμενο των συζητήσεών μας σήμερα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Σταθεροποίησης ε, θα συγκροτηθεί και θα είναι ένα κομμάτι του μοσαϊκού ε, της ε, πιο ευμερούσας ε, Ευρώπης. Θα έχουμε καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση, θα λειτουργούν καλύτερα χρηματοπιστωτικές αγορές. Με αυτές τις έξι προτάσεις που έχουμε αναχείρας εκινήσαμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι του παζλ μόλις περατωθεί. Με αυτά και με τη σημερινή μας συζήτηση ευελπιστώ το Μάρτιν να ληφθεί μια θετική απόφαση. Πάντως έχουμε στείλει σαφή μηνύματα προ όλου όσου είχαν, είχαν στοιχηματίσει κατά του ευρώ. Αν στοιχηματίσετε κατά του ευρώ, του λέμε, θα χάσετε τα λεφτά σα. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα και ε, θα έπρεπε να το μεταφέρουμε. Ε, στους σκεπτικιστές. Είναι κέρια σημασία η απόφαση που θα ληφθεί το Μάρτιο. Βλέπω ότι για τους βουλευτές είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρηθούν απολύτως οι αρμοδιότητες ε, της Ένωσης και να ε, σεβαστούμε το ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου της Ένωσης. Προφανέστατα θα μεριμνήσουμε ώστε όλα, όλες οι διατάξεις να είναι με το κοινοτικό κεκτημένο. Σχετικά με το μηχανισμό, πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μία συνέπεια με το συνολικότερο πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης κυρίως όταν μιλάμε για τον συντονισμό ε, και την παρακολούθηση των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερως δε των κρατών μελών που, είναι, ε, που ανήκουν στην ζώνη του ευρώ. Κάποιοι εξέφρασαν ε, ανησυχίε ε, ότι θέλουν να οικοδομήσουν μια Ευρώπη δύο και περισσότερων ταχυτήτων. Είναι σαφέστατη η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού παρότι η πρωτεύουσα ευθύνη ε, για το ενιαίο νόμισμα ανήκει στα κράτη-μέλη τη ζώνη ευρώ. Είναι σαφέστατο ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό ο μηχανισμό και σε άλλα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ και για να επιτύχουμε μεγαλύτερη οικονομική σύγκληση καλό θα ήταν να συμμετάσχουν και τα 27 κράτη-μέλη. Η προϊούσα διαδικασία λοιπόν δείχνει ότι θα αναλάβουν λένε και πιο δραστήριο ρόλο και οι ίδιες οι χρηματοπιστωτικές αγορές για να ενισχυθεί η συνεργασία μας στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο μόνο θα καταστήσουμε ε, ισχυρότερη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερους τους ε, συνεισηγητές, ε, τον κύριο Γκολτιέρη και τον κύριο Μπρόκ, για τις προτάσεις, τις ιδέες που κατέθεσαν τις, και τους ευχαριστούμε για τις διαβουλεύσεις, μόνιμες διαβουλεύσεις που έχουμε μαζί τους εργαζόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο Καταλήξατε στην έκθεση που αναμένεται γέρος να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ε, βεβαίως από το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τελευταία παρατήρηση προς τον κύριο Τζο Χίγκινς ε, από την Ιρλανδία. Ορθότατα ε, η παρέθεσε τον Επίτροπο ε, Ρεν ε, και ο οποίος είπε ότι με την Ιρλανδία ως χώρα και όχι ως κυβέρνηση ε, συνάψαμε τη συμφωνία και ευελπιστούμε ότι θα τηρηθεί η συμφωνία φωτέρων των πλευρών. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προβλημάτων με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ιρλανδία και ελπίζουμε αμελητή να ανακάμψει η Ιρλανδία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της Ιρλανδίας και ελπίζουμε να επιστρέψει η ανάπτυξη και η ευημερία στην Ιρλανδία το ταχύτερο δυνατόν χάρη σε αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πέρα στη συζήτηση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η κατάσταση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος σε θέματα ασύλου μετά την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.